Uh, good afternoon απόγευμα λοιπόν. Ας αρχίσουμε. Πρώτο θέμα έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ο εισηγητής του θέματος TDI ζήτησε να κάνουμε την ψηφοφορία για το σημείο 11 της ημερήσιας διάταξης στο τέλος του απογεύματος. Μήπως υπάρχει αντίρρηση. Αν όχι, το δεχόμαστε. Προχωρούμε. Λοιπόν, σημείο 2. Έγκριση των πρακτικών των παλιότερων συνεδριάσεων του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου. Θα θεωρηθούν εγκεκριμένα τα πρακτικά αν δεν υπάρξουν ενστάσεις, αντιρρήσεις μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Σημείο 3 τώρα, Ανακοινώση του Προέδρου. ε, να σας ειδοποιήσω ότι περνάει από το διαδίκτυο web streaming η σημερινή συνεδρίαση εκτός βεβαίως από τη συνεδρία των συντονιστών που δεν μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Τώρα, ε, ειδήσει Μερκοσούρ, η Ευρωπαϊκή Ένωση κοινοποίησε ότι μετά η 19ης ε, Δεκεμβρίου η Βραζιλία ε, έκανε επίση κάποιες κοινοποίησεις έδωσε ορισμένες, ε, ορισμένα νέα για το τομέα At the same Ζήτησε διαβουλεύσεις για ορισμένους τομείς και οι ε, Αργεντινοί ζήτησε να συζητηθούν τα μέτρα αντι-dumping της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Τετάρτη 22 Ιανουαρίου μεθαύριο λοιπόν θα γίνει συνάντηση για θέματα Μερκοσούρ Βιετνάμ γιατί... Στις 13 και 17 Ιανουαρίου έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες με συνεδρίαση για την ενδεχόμενη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου και οι διαβουλεύσεις πήγαν καλά. Το επόμενο, ο έβδομος γύρος θα λάβει χώρα μέσα Μαρτίου στο Βιετνάμ. Τώρα PA και Trade Promotion Authority αυτό είναι το TPA σχετικά έγιναν κάποιες πρόοδοι για τα πρότυπα ε, συζητήθηκαν συζητήθηκε το θέμα της διαφάνειας διαβουλεύσεων συμμετοχή του Κογκρέσου στις διαβουλεύσεις καταλαβαίνετε ότι είναι ε, αμερικάνικη συνήθεια αυτή η συμμετοχή του Κοινοβουλίου αν θέλετε στις διαπραγματεύσεις του εμπορικών συμφωνιών δεν ξέρω αν θέλουμε να ε, συμμετάσχει το Κογκρέσο σε αυτές τις διαβουλεύσεις για το, και για το τίπιτ τότε θα έπρεπε να συμμετάσχει το Κογκρέσο θα πρέπει να το δούμε για το Σιγκαπούρη η Καναδά ΣΥΤΕΠ δεν υπάρχουν πολλές καινούργιες ειδήσει για να σας ενημερώσω δεν είναι έτοιμη η καινούργια συμφωνία ΣΥΤΕΠ Ας προχωρήσουμε όμως στο σημείο 4, ουσιαστικό θέμα της ημερήσιας διάταξης. Έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος, τον κύριο Νότι Μηταράκη, που είναι υπεύθυνο, αρμόδιος, μεταξύ άλλων, για τις εξαγωγές και τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις στην ε, ελληνική κυβέρνηση. Εκπροσωπεί την ενεργεία προεδρία του Συμβουλίου θα είναι ο συνομιλητής μας στο Συμβούλιο για τους επόμενους έξι μήνες. Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκεται εδώ ο κύριος Μηταράκης και η ομάδα του και έχουμε μαζί μας και το νέο ε, αρμόδιο αν θέλετε της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας μετά από τον θάνατο σε τροχαίο του προηγουμένου εκπροσώπου της Ελλάδας ε, είναι μαζί μας η κυρία η διάδοχος χαίρομαι λοιπόν που είστε εδώ συνάντησα τον κύριο Μηταράκη και εδώ και στην Αθήνα κατά την επίσκεψή μου στην Ελλάδα ήταν πραγματικά πολύ ευχάριστη η συνάντηση μαζί του και θα δείτε τώρα που θα σας μιλήσει έχει σαφέστατες απόψεις ε, για το τι θα γίνει κατά τη διάρκεια της Προεδρίας. Λοιπόν, χαιρόμαστε που είστε εδώ. Βεβαίως ε, η παρουσίαση που θα μας κάνει ο κύριος Υπουργό τώρα είναι η συνείδηση παρουσίαση που γίνεται στην αρχή της κάθε προεδρίας όπου πραγματικά ε, παρουσιάζεται το πρόγραμμα της προεδρίας και οι προτεραιότητες. Εδώ θα μιλήσουμε για τις προτεραιότητες εμπορικές και επενδυτικές. Κύριε Υπουργέ, χαιρόμαστε που είστε εδώ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, Επιτρέψτε μου με την ιδιότητα επίσης του βουλευτού του Ελληνικού Εθνικού Κοινοβουλίου να πω κυρίε και κύριοι συνάδελφοι. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, τιμή και συγκίνηση που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας για τους επόμενους έξι μήνες και να ανταλλάξω από αυτόν απόψει μαζί σα. Για την ε, Προεδρία είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκφράζει τους λαούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στους επόμενους έξι μήνες, κύριε Πρόεδρε, όπως έχουμε ήδη συζητήσει στις διμερείς μας επαφές, η Προεδρία θα καταστήσει κάθε δυνατή προσπάθεια να έχει ένα ανοιχτό διάλογο με το Ευρωκοινοβούλιο. Η συνεργασία ειδικά με την Επιτροπή σας στην ΙΝΤΑ είναι η συνέχεια μιας συνεργασίας που έχουμε εγκαινιάσει ήδη με επιτυχία. Καθώς με τον καθηγητή τον κύριο Μορέιρα αλλά και τα άλλα μέλη της Επιτροπής σας είχαμε τη δυνατότητα καταρχήν να συνεργαστούμε στενά κατά την πρόσφατη σύνοδο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου στην Ινδονησία, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετείχε με μια σημαντική αποστολή. Αλλά και στην Αθήνα είχαμε πρόσφατα την ευκαιρία να σας υποδεχτούμε μαζί με τον κύριο Καζάκ και να συζητήσουμε τρόπους συντονισμού της δράσης μας και για γενικότερα και για ειδικότερα θέματα γιατί πέρα από οποιασδήποτε ιδεολογικές διαφορές όλοι προσπαθούμε για μια καλύτερη Ευρώπη για τους λαούς της και για τους πολίτες της. Και βεβαίως μέσα σε αυτή την Ευρώπη τα θέματα του εμπορίου έχουν κομβικό ρόλο. Γιατί η επιτυχής κατάληξη των συμφωνιών που συζητούμε θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ενίσχυση της ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που απασχολούν σήμερα όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Πώς θα επιτύχουμε ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης και πώς θα πετύχουμε τη μείωση της ανεργίας που μας βασανίζει όλους. Και σε αυτό ο ρόλος του ελεύθερου διεθνούς εμπορίου ε, παίζει καταλητικό ρόλο. Οι προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας σε αυτό το διάστημα συγκεντρώνονται γύρω από τέσσερις πυλώνες δράσης. Η πρώτη προτεραιότητα είναι η αναχώρα κάθετες διμερείς διαπραγματεύσεις. Η Ελλάδα θα προσπαθήσει να διευκολύνει το διάλογο των κρατών μελών μεταξύ τους και με το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο τον άρτιο συντονισμό της Ευρωπαϊκής Διαπραγματευτικής Στρατηγικής σε ό,τι αφορά στις διμερείς εμπορικές συμφωνίες. Το εν λόγω θέμα είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην περίπτωση συμφωνιών μεικτή αρμοδιότητα, δηλαδή συμφωνιών που άπτονται θεμάτων εκτό τη κοινή εμπορική πολιτική, το οποίο αφορά την πλειονότητα των διμερών συμφωνιών προς διαπραγμάτευση. Πρώτη προτεραιότητα οι διαπραγματεύσεις για τη Διατλαντική Εμπορική και Επενδυτική Εταιρική Σχέση, TTIP. Αναμένουμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τους γύρους διαπραγματεύσεων που έχουν ήδη ολοκληρωθεί την ανταλλαγή προσφορών που θα λάβει χώρα στις 10 Φεβρουαρίου και μία εβδομάδα μετά την απογραφή πολιτικής που θα λάβει χώρα ανάμεσα στον Ευρωπαίο Επίτροπο, στον κύριο Τιγκούχτ και στον Αμερικάνο High Trade Representative, τον κύριο Φρόμεν. Στο άτυπο Συμβούλιο της Αθήνας, στις 27 και 28 Φεβρουαρίου, θα δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συζήτηση πάνω στη Συμφωνία TTIP. Στο πρόγευμα εργασίας θα δώσουμε τη δυνατότητα σε εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας και της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών να παρουσιάσουν στα μέλη του Συμβουλίου και στον καθηγητή τον κύριο Μορέιρα που θα είναι ιδιαίτερη τιμή να προσκαλέσουμε στο άτυπο Συμβούλιο της Αθήνας τις απόψεις της αγοράς για αυτή τη συμφωνία. Και μετά, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών, να συζητήσουμε τις εξελίξεις και να δούμε τις θέσεις των κρατών μελών. Δεύτερο σημαντική προτεραιότητα για μας είναι η ολοκλήρωση του εμπορικού συμφώνου Καναδά-Ευρωπαϊκής Ένωσης, ΣΕΤΑ. Όπως γνωρίζουμε, οι τεχνικές και νομικές του πτυχές είναι υπό Μόλι ολοκληρωθούν η διαδικασία διαπραγματευση και η νομική εξέταση, τα μέρη θα είναι έτοιμα να προχωρήσουν στη μονογραφή τη συμφωνία. Ευελπιστούμε να υπάρξουν εξελίξει κατά τη διάρκεια τη ελληνική Προεδρία. Τρίτη προτεραιότητα στον άξονα διμερών συμφωνιών είναι οι διαπραγματεύσει Ευρωπαϊκή Ένωση Ιαπωνία για Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται να υποβάλει έκθεση τον Απρίλιο σχετικά με την εφαρμογή των δεσμεύσεων που ανέλαβε η Ιαπωνία για την εξάλληψη των μη δασμολογικών εμποδίων, καθώ και την ανάγκη για αυξημένη πρόσβαση στου δημόσιους διαγωνισμού προμηθειών για του σιδηροδρόμου και για τι αστικέ συγκοινωνίε. Ανάλογα με την πρόοδο που θα σημειωθεί, το Συμβούλιο θα συζητήσει κατά τη σύνοδό του στι 8 Μαου στι Βρυξέλλε κατά πόσο χρειάζεται να γίνει μια επανεξέταση των ειδικιών που έχουν δοθεί. Τέταρτον, θα επιδιώξουμε, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με Κίνα, τις χώρες τη Μεσογείου και τις χώρες του κόλπου, να προωθήσουμε τις διμερείς συμφωνίες που ήδη συζητούνται. Αποτελούν οι χώρες αυτές μείζονες εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην παγκόσμια αγορά. Ειδικά για τις χώρες του Μεσογείου, να τονίσω ότι μια προτεραιότητα της ελληνικής προεδρίας, όχι στο Συμβούλιο Εξωτερικού Εμπορίου αλλά κεντρικές προτεραιότητες, οι τέσσερις κεντρικές προτεραιότητες είναι και η ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεωρούμε ότι στην κατεύθυνση αυτή η βελτίωση των εμπορικών σχέσεων της Ένωσης με τις χώρες οι οποίες συνορεύουν με εμάς συμβάλλει θετικά σε αυτή την παράμετρο. Τέλος, αναφορικά με τις χώρες της Μερκονσούρ γνωρίζουμε ότι έχουν πραγματοποιηθεί ως σήμερα 9 διαπραγματευτικοί γύροι και ο τελευταίο τον Οκτώβριο του 2012. Οι διαπραγματεύσεις με τις χώρες αυτές έχουν επικεντρωθεί στο κομμάτι της συμφωνίας που αφορεί τους κανόνες και τα δύο μέρη εργάζονται προς την κατεύθυνση της προετοιμασίας των προσφορών για πρόσβαση στην αγορά. Δεν έχει όπως γνωρίζετε καθοριστεί ακόμα ημερομηνία υποβολής των ελόγων προσφορών παρότι υπάρχουν πλέον θετικές ενδείξεις ιδιαίτερα από την πλευρά της Βραζιλίας. Αυτό είναι ο πρώτος πυλώνας προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας. Ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται σε οριζόντιες προτεραιότητες και θα αναφερθώ σε δύο. Πρώτον, η ανάγκη για αυξημένη προστασία των προϊόντων προστατευμένης γεωγραφικής ένδειξης και προστατευμένων προϊόντων ονομασίας προέλευσης. Η αυξημένη προστασία των υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έχουν πιστοποιηθεί ως ΠΟΠ και ως προϊόντα ΠΓΕ θα παραμείνουν προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά το όλο το πνεύμα των διμερών εμπορικών διαπραγματεύσεων, καθώς συνδέεται στενά με τη διαθροτική μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Γεωργίας, καθώς και με την ανάγκη επιτυχούς πρόσβασης των παραδοσιακών υψηλής προστιθέμενης αξίας ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Σημειώνουμε ότι στη συζήτηση του TTIP το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή σας, με το δήλωση του Προέδρου, είχε πει πολύ συγκεκριμένα ότι χωρίς συμφωνία για τα προϊόντα γεωγραφικής ένδειξης και τα προϊόντα POP δεν είναι δυνατόν να επέλθει συμφωνία. No GIs, no deal, όπως είχε πει ο Πρόεδρος ο κ. Μορέιρα. Η Ελληνική Προεδρία στο άτυπο Συμβούλιο της Αθήνας θα παρουσιάσει και νέες σκέψεις κατά πόσο μπορούμε να ενισχύσουμε το μηχανισμό προστασίας αυτών των προϊόντων. Θα θέσουμε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα κατά πόσο χωρίς αυτό να αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σήμερα διαπραγματευόμαστε στις διασύνες μας συμφωνίες αυτά τα προϊόντα, κατά πόσο η Ευρώπη θα έπρεπε να κατοχυρώσει και με το αγγλοσαξονικό νομικό σύστημα ένα ευρωπαϊκό σήμα, trademark, να το γράψει, να το κατοχυρώσει διεθνώς και με το οποίο να πιστοποιούνται τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Ένα trademark το οποίο θα αντανακλά τα νομοθετικά συστήματα κρατών που σήμερα δεν έχουν αποδεχτεί την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα ΠΟΠ. Ένα δεύτερο θέμα πρέπει να συζητήσουμε είναι κατά πόσο σε διμερείς συμφωνίες της Ένωσης που μιλάμε για προϊόντα ΠΟΠ ζητούνται μεταβατικές ή άλλες διατάξεις από χώρες τα οποία όμως δεν αφοράνε δικιά τους παραγωγή και κατά πόσο μπορούν δηλαδή οι Ευρωπαίοι παραγωγοί όλοι να συμβάλλουμε και εμείς στην προστασία των δικών μα σημάτων ΠΟΠ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, ως προς τις οριζόντες προτεραιότητες, να αναφέρω τις ναυτιλιακές πλευρές της εμπορικής πολιτικής. Η τέταρτη κεντρική προτεραιότητα της Ελλάδος ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ναυτιλία, η γαλάζια ανάπτυξη. Να υπογραμμίσω ότι το θαλάσσιο εμπόριο αποτελεί σήμερα το 90% μεταξύ του συνολικού, εμπορίου, του, συνολικού εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών και το 40% του ενδοευρωπαϊκού εμπορίου. Άρα η ναυτιλία είναι καθοριστικός παράγοντας για την οικονομική ανάπτυξη και ευμάρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και εγγυητή για την ομαλή ροή των ευρωπαϊκών εισαγωγών και εξαγωγών παγκοσμίω. Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, η ελληνική προεδρία θα εργαστεί για να διασφαλίσει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών θα συμπεριλαμβάνουν τυποποιημένα κείμενα περί θαλάσσιων μεταφορών και ειδικά περί απελευθέρωσης των λαυτιλιακών υπηρεσιών. Πηγαίνω στον τρίτο πυλώνα, στις πολυμερείς συμφωνίες. Ως προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, στον απόϊχο της θετικής συμφωνίας του Παλί, η προσοχή τώρα του Παγκόσμιου Οργανισμού θα εστιαστεί σε θέματα που δεν επιλύθηκαν στην Ινδονησία, καθώς και σε άλλα θέματα της αναπτυχιακής ατζέντα της Ντόχα. Από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό συνεπάγεται την ανάγκη πραγματοποίησης ενός σοβαρού απολογισμού του αποτελέσματος του Μπαλή από το Συμβούλιο, αλλά και τη διεξαγωγή ενός στρατηγικού διαλόγου για την κατεύθυνση στην οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει να στραφεί ο ΠΟΕ. Κατά το άτυπο δείπνο των Υπουργών Εξωτερικού Εμπορίου στην Αθήνα στις 27 Φεβρουαρίου, στο οποίο όπως τόνισα θα είναι παρόν και ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Μορέιρα, θα συζητήσουμε την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τον Παλί. Να τονίσω επίσης στο θέμα των περιμερών συμφωνιών τη σημασία που δίνουμε σε μη δασμολογικά εμπόδια Μεταξύ των προβλημάτων που καλούμεθα να επιλύσουμε στην περίοδο μετά τον Παλή είναι η υιοθέτηση μέτρων που θα βελτιώσουν την πρόσβαση στην αγορά. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ένα από τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν είναι η απάλληψη των μη δασκολογικών εμποδίων. Το θέμα αποτελεί σίγουρα προτεραιότητα, δεδομένου ότι μεγάλο μέρο των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει στι εξαγωγικέ του δραστηριότητε συνδέονται με αυτά τα εμπόδια. Τα κύρια θύματα αυτής της κατάστασης είναι κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες ωστόσο αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε αυτά τα πλαίσια ενθαρρύνεται η συμβολή των κρατών μελών, ειδικά με τη μορφή πληροφόρησης και έρευνας που γνωρίζουμε ότι γίνεται, που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ποσοτικοποίηση του βαθμού στο οποίο αυτά τα εμπόδια εμποδίζουν τις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Τέταρτη προτεραιότητα, ιδιαίτερα σημαντική, παρότι την αναφέρω απλώς φωνολογικά τέταρτη, αλλά για μας είναι κρίσιμη προτεραιότητα, είναι να λειτουργήσουμε ως αξιόπιστος μεσολαβητής στους τριλόγους, οι οποίοι έχουν να κάνουν με την νομοθετική εργασία του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ο στόχος είναι να προωθήσουμε φακέλους και να μπορέσουμε να κλείσουμε θέματα που εκκρεμούν. Βασική αρχή της ελληνικής προεδρίας, όπως την καθόρισε και ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο κ. Αντώνης Σαμαράς, είναι να μπορέσουμε λόγω του γεγονότος ότι το Ευρωπαϊκό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώνει τη θητεία του σε αυτό το συντομότερο από συνήθω εξάμεινο διάστημα να, να προσπαθήσουμε όπου αυτό είναι δυνατό να κλείσουμε διαλόγους οι οποίοι, οι οποίοι ακόμα εκκρεμούν. Ως προς τον κανονισμό χρηματοδοτικής ευθύνης. Ως Προεδρία είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε με γρήγορα βήματα τη διαδικασία της υιοθέτησης. Και αυτό διότι αναγνωρίζουμε πρώτον την ανάγκη οι συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιλαμβάνουν θέματα προστασίας των επενδύσεων να συμπεριλαμβάνουν και το θέμα της επίλυσης διαφορών μεταξύ κράτους και επενδυτών. Και δεύτερον, αναγνωρίζουμε την ανάγκη καθορισμού και κατανομής της ευθύνης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών στις συγκεκριμένε περιπτώσεις. Όπως γνωρίζετε αυτή η συζήτηση αφορά, χωρίς να θέλω να μπω τεχνικά θέματα, τα άρθρα 8 και 9 που σχετίζονται με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία από τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλάβει την υπεράσπιση μιας υπόθεσης αποσπώντας της από το κράτο μέλος. Έχει δοθεί ένα κείμενο της Επιτροπής στα κράτη-μέλη στις 15 Ιανουαρίου και το Trade Policy Committee, Service και Investment δεν μπορούσε να το συζητήσει εκείνη την ημέρα διότι δεν είχαν προλάβει οι αντιπροσωπείες να το διαβάσουν αλλά θα συζητηθεί κατά την επόμενη συνεδρία της Επιτροπής στις 29 Ιανουαρίου. Επί της ουσίας, η θέση μας είναι ότι η συγκεκριμένη πρόταση κινείται στη σωστή κατεύθυνση και αντανακλά ειλικρινή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να προσεγγίσει τις θέσεις των κρατών μελών. Είμαστε ήδη σε επαφή με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή για να προσδιορίσουμε επακριβώς τις ημερομηνίες για τον επόμενο τρίλογο, επιδιώκοντας σε κάθε περίπτωση να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση ώστε να μπορέσουμε να προλάβουμε να επιτευχθεί συμφωνία αν τελικά το τελικό κείμενο ανταποκρίνεται στις απαιτήσει όλων των εμπλεκομένων μερών στη διάρκεια αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Δεύτερος πολύ σημαντική πρωτοβουλία είναι η οδηγία για την εφαρμογή και επιβολή εμπορικών κανόνων, το Trade Enforcement. Σχετικά με το συγκεκριμένο κανονισμό σημειώνουμε τη σημασία που έχει την ισχυροποίηση τη θέση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν διαπραγματεύεται διεθνεί εμπορικέ συμφωνίε. Και βεβαίω να αντιδρά με τόπο ταχύ και όχι μετά από χρονοβόρε διαδικασίε συναπόφαση. Στόχο μα είναι να επιτύχουμε μια συμβιβαστική συμφωνία αποδεχτεί και από τα τρία όργανα, λαμβάνοντα υπόψη την προθεσμία 12-13 Φεβρουαρίου για να υιοθετηθεί το ντοσιέ από την Επιτροπή σα. Παρά την πολυπλοκότητα του θέματος, Πιστεύουμε ότι έχει γίνει σημαντική πρόοδος, ειδικά με την εξέταση της συμπερίληψης των υπηρεσιών σε μια μελλοντική επανεξέταση. Εστιάζουμε τις προσπάθειές μας στην εξέβρεση κοινού τόπου, σχετικά πρώτον με τη διαδικασία προσδιορισμού των συμβαλόμενων αρχών ή νομικών οντοτήτων στον τομέα των δημόσιων συμβάσεων και δεύτερον στην ανταλλαγή πληροφορίας μεταξύ των οργάνων υπάρχουν άλλε δύο νομοθετικέ πρωτοβουλίες. Η πρωτοβουλία των Διεθνών Δημοσίων Συμβάσεων και η θετική σας ψήφος στι 15 Ιανουαρίου έδωσε το πράσινο φω και είμαστε έτοιμοι για να ξεκινήσει ο τρίλογος. Θα προσπαθήσουμε σε αυτή την, σε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία να γεφυρώσουμε τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών. Τέταρτον, αναφορικά με τον εξυγχρονισμό εργαλείων εμπορικής άμυνας, αντι-dumping, αντι-subsidy measures. Εδώ οι διαφορέ υπάρχουν τόσο μεταξύ των οργάνων όσο και εντό του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι ένα δύσκολο φάκελο. Ω Προεδρία φιλοδοξούμε να συμβάλλουμε στον εξυγχρονισμό χωρίς βεβαίως να χαθεί η αποτελεσματικότητα των εν λόγω εργαλείων. Αναμένουμε το αποτέλεσμα τη αυριανή σα ψηφοφορία για να προχωρήσουμε. Σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη θα κάνουμε τι κινήσει μα ώστε να επιτύχουμε τη σχετική εντολή για να προχωρήσουμε, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη και το ασφιχτικό χρονικό πλαίσιο που υφίσταται. Είναι προφανές, κυρίε και κύριοι συνάδελφοι, ότι έχουμε μπροστά μας ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Το θετικό στοιχείο είναι το πνεύμα συνεργασίας που βλέπω σε όλα τα άργανα παρά τη διαφορά αντιλήψεων που υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις. Το οποίο είναι στοιχείο της δημοκρατίας και του πλουραλισμού που υπάρχει στην Ευρώπη. Και είμαι πεπισμένος ότι με τη βοήθεια όλη, όλων, με τη λήξη της Προεδρίας, θα είμαστε θέση να παρουσιάσουμε πρόοδο και επιτεύγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδιαίτερα τιμητική πρόσκληση που μου απευθύνεται σήμερα, κύριε Πρόεδρε, να απευθυνθώ στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Ξεκινούμε τις ερωτήσεις ή παρατηρήσεις. Ο κ. Καζάκα από τους Φιλελεύθερους. Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, θα ήθελα καταρχάς να σας καλωσορίσω εκ νέου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όπως και ο πρόεδρος ε, της Επιτροπής ανέφερε, είχαμε την δυνατότητα να σας συναντήσουμε κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στην Αθήνα στο τέλος του 2013. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε μια ανταλλαγή απόψεων αρκετά λεπτομεριακή θα έλεγα για τις προτεραιότητες της ελληνικής προεδρίας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι μας, είχε εντυπωσιάσει πολύ η φιλοδοξία και ο ενθουσιασμός που η ελληνική προεδρία είχε εκδηλώσει για θέματα εξωτερικού εμπορίου. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ωστόσο ότι η διάρκεια της προεδρίας σας θα είναι βραχύτερη από ό,τι συνήθως λόγω των ευρωεκλογών του Μαΐου έχετε δύο-τρεις μήνες μόνο για να, για να δράσετε. Κάτι που απαιτεί μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση από πλευρά σας καθώς και μια αναζήτηση εταίρων που θα συμμερίζονται τις απόψεις σας για να αντιμετωπίσετε τις προκλήσεις αυτές. Θα ήθελα να θέσω μια σειρά ερωτημάτων μετά την παρέμβασή σας. Είπατε ότι τον Απρίλιο θα προχωρήσετε σε μια απογραφή της κατάστασης ε, σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ένωσης και Ιαπωνίας. Είμαι εισηγητής στο Κοινοβούλιο για τον ε, φάκελο αυτό και θέλω να σας ε, ρωτήσω την άποψή σας. Είστε αισιόδοξο ως προς τα αποτελέσματα της απογραφής αυτής της κατάστασης. Μέχρι τότε θα έχουμε λόγους για να ελπίζουμε ότι θα υπάρξουν λύσεις ως προς την απουσία των μη δασμολογικών εμποδίων και την πρόσβαση των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Ιδίως δε στις κρατικές προμήθειες για θέματα σιδηροδρομικά. Η απογραφή θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε ταχύτερα στις διαπραγματεύσεις. Μετά, έκθεση Κάσπαρη για την πρόσβαση στις ε, κρατικές προμήθειες, έκθεση που ψηφίστηκε στην προηγούμενη Ολομέλεια. Ε, ξέρετε καλύτερα από μένα ότι υπάρχουν επιφυλάξεις και διαφορές στο εσωτερικό του Συμβουλίου. Είναι σοβαρές αυτές οι διαφορές. Πιστεύετε ότι ο συμβιβασμός που θα πετύχουμε στην Ένωση θα αποτελεί επαρκώς στέρεη βάση για να υπάρξει συμφωνία στο Συμβούλιο που έχει επιφυλάξει και να μπορέσουμε να έχουμε μια κοινή θέση για τον κανονισμό αυτό. Στην, η επίσκεψή σας εδώ συμπίπτει με μια άλλη σημαντική επίσκεψη του Τούρκου Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας της χώρας που είναι εδώ στις Βρεξέλλες σε επίσημη επίσκεψη. Περιμένουμε συζητήσεις για τις διμερείς σχέσεις στον τομέα του εμπορίου και της Τελωνιακή Ενώσεως. Πιστεύετε ότι κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας ε, θα μπορέσει να δοθεί μια όθηση στην λειτουργία της Τελωνιακής Ένωσης μεταξύ ΕΕ και Τουρκίας για να επιληθούν τα εκκρεμή ζητήματα, ιδίως ε, αυτά που αφορούν την ισότιμη αντιμετώπιση της Τουρκίας κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων για την ελεύθερη κυκλοφορία με τρίτες χώρες. Ευχαριστώ και καλή επιτυχία. Next, uh, Paul Murphy, United European Left. No, Scholz. Ah, no. Ο επόμενος. My indication was Paul Murphy. Now I have Helmut Scholz. I... Κύριος Murphy. Ο... ο... Κύριε Σούλτ, δεν ξέρω αν θέλει ο Πολ Μέρφυ το λόγο. Ευχαρίστως. Θα ήθελα, εν περιπτώσει, εγώ να ευχαριστήσω τον Ευρωπουργό για την λεπτομερέστατη και εκτενή παρουσίαση των στόχων της ε, ελληνικής προεδρίας. Ε, μας ανέφερε ε, πάρα πολλά θέματα τα οποία θα απασχολήσουν την Προεδρία. Ε, γι' αυτό έχω ορισμένα ερωτήματα να θέσω. Μιλήσατε για προτεραιότητες και προ... αρκετά ψηλή προτεραιότητα ε, μας αναφέρατε ποια θέματα έχουν ερώτηση λοιπόν πώς βλέπετε την κατάσταση στο Συμβούλιο ε, πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσει το Συμβούλιο ε, στον επόμενο γύρο βάσει των εμπειριών των προηγούμενων γύρων αυτοί που έχουν παρακολουθήσει τις διαβουλεύσεις ε, ξέρουν πολύ καλά ότι τα πράγματα πάνε είναι μάλλον δύσκολο αλλά εσείς πώς πιστεύετε ότι θα αντιδράσει το Συμβούλιο και πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσε να συνεργαστούν καλύτερα ε, το Συμβούλιο με το Κοινοβούλιο ως δύο ε, κλάδι του νομοθε... της νομοθετικής εξουσίας αν θέλετε στα ευρωπαϊκά όργανα για το θέμα των προτύπων ή ε, για ιδιαίτερα στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Ξέρετε πολύ καλά ότι ε, έχουμε ε, κάποια, βρισκόμαστε σε ένα ψηλό επίπεδο προτύπων ε, σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου. Τα πρότυπά μας είναι αρκετά ψηλά. Αν θέλετε τα standards μας τι πιστεύετε ότι θα γίνει εκεί. Δεύτερο θέμα. Είπατε ότι μεταξύ των οριζόντιων θεμάτων θα α, περιλαμβάνονται όχι μόνο το τι το TTIP αλλά και διμερείς συμφωνίες που, όπου έχουμε και την συμφωνία με την Κίνα και τα λοιπά ε, πώς φαντάζεστε πώς είναι η κατάσταση για τα θέματα αυτά στο Συμβούλιο πιστεύετε ότι θα υπάρξει πρόοδος ή θα παραμείνουν τα προβλήματα που ξέρουμε ότι υπάρχουν στο Συμβούλιο αυτό αυτή τη στιγμή. Τώρα επειδή είμαι εισηγητή για τα θέματα με την Κίνα να πω ότι το Συμβούλιο εδώ ε, όρισε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που θα ήθελε να ακολουθήσει και όρισε, όρισε και ορισμένα σοβαρά θέματα για την αμοιβαία πρόσβαση στην αγορά παραδείγματος χάρη. Και εδώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω η Ελλάδα σαν προεδρεύων του Συμβουλίου αυτή τη στιγμή πώς θα αντιμετωπίσει το θέμα της Κίνας. Ε, ξέρουμε πολύ καλά ότι οι Κινέζοι εκμεταλλεύονται μια κάποια οικονομική κατάσταση που υπάρχει εδώ αλλά θα ήθελα πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Τώρα για την συμφωνία ΣΕΤΕΠ να ρωτήσω το εξής. Το Συμβούλιο έχει συνέστηση ότι ορισμένα κεφάλαια κλείσανε. Πώς πιέζει η Κομισιόν ή το Συμβουλίο των Κομισιόν να ξανανοίξουν να ανοίξουν ορισμένα κεφάλαια για να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια. Και κάτι τι άλλο κλείνοντας μιλήσατε για την πολιτική γειτονίας. για την ασφάλεια, για τη σταθερότητα ενδιαφερόμαστε και εμείς που είμαστε που ασχολούμεθα με τα εμπορικά πράγματα ε, στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας ε, εσείς πώς βλέπετε να κινούνται τα πράγματα εδώ ε, στη Μεσόγειο πιο συγκεκριμένα και στη Μέση Ανατολή αλλά ειδικότερα στη Μεσόγειο ευχαριστώ uh, για συντηρητικούς ο συνάδελφος κύριος Έπινγκ. Μία ερώτηση προς τον Υπουργό θέλω. Μπορεί να μας διευκρινίσει η Προεδρία αν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της προβλέπεται σύνοδος κορυφής με την Ρωσική Ομοσπονδία για να επανενεργοποιηθούν οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία πλαίσιο ένωσης Ρωσίας και πώς πιστεύει ο υπουργό ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της Ουκρανίας διότι οι διαπραγματεύσεις ε, δεν οδήγησαν σε αποτέλεσμα μεταξύ άλλων λόγω της ρωσικής πίεσης πώς θα θέσουμε στο σωστό δρόμο τις σχέσεις μας με την Ουκρανία ξανά. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, είναι ο πρώτος γύρος απαντήσεων, θα υπάρξει και δεύτερος ε, ερωτήσεων. Παρακαλώ, αν θέλετε να απαντήσετε τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Για τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις τις οποίες μου έχετε απευθύνει. Ε, με τον κύριο Καζάκ πράγματι είχαμε τη δυνατότητα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας κατά την επίσκεψη της Επιτροπής στην Αθήνα και σας ευχαριστώ και άλλη μια φορά για τη συμμετοχή σας ε, τον προηγούμενο μήνα. Ως αναφορικά με τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Ιαπωνίας, θέλω να είμαι αισιόδοξο ότι θα μπορέσει να υπάρξει μια θετική εξέλιξη που να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 8 Μαΐου να θεωρήσει ότι οι διαπραγματεύσεις οδηγούνται είναι σε καλό δρόμο. Βέβαια, είμαστε υποχρεωμένοι να αναθεωρήσουμε τη θέση μας αν τελικά η, η πραγματικότητα είναι χειρότερη από τις αρχικές μας θετικές προσδοκίες. Είναι σημαντικό η εμπορική συμφωνία αυτή να ανοίγει αγορές της Ιαπωνίας για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ο στόχος των διμερών συμφωνιών είναι πάντα η δημιουργία τελικά θέσεων εργασίας και να ανοίγουμε αγορές. Και αν μια συμφωνία δεν μπορεί να το πετύχει αυτό, είναι κάτι που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Αναφορικά με την έκθεση Κασπάρη, αναφέρθηκα ως προς το θέμα του public procurement, ως προς το θέμα του τριλόγου, ότι ακόμα υπάρχουν σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Είναι κάτι που συνεχίζουμε να συζητούμε και η ελληνική προεδρία ως προεδρεύουσα χώρα ο ρόλος της είναι να, βοηθήσει στην εξέβρεση κοινού εδάφους όπου αυτό βέβαια είναι εφικτό. Η διάρκεια της Προεδρίας παραμένει εξάμηνη βέβαια, αλλά η διάρκειά μας ε, για να λειτουργήσουμε ε, στους τριλόγους είναι περιορισμένη, αλλά θα προσπαθήσουμε σε αυτό το σύντομο διάστημα να κάνουμε ό,τι είναι εφικτό. Αναφερθήκατε συγκεκριμένα για το θέμα της Τουρκίας και σας θυμίζω ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας αποτελεί και για τη χώρα μου μια σημαντική προτεραιότητα. Και παραμένει μια σημαντική προτεραιότητα. Η σταθερότητα, η πολιτική, η οικονομική ανάπτυξη της Τουρκίας είναι προς όφελος και των διμερών οικονομικών σχέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά θα λειτουργήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση έχοντας και τις πολύ καλές σχέσεις γειτονίας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Ως προς, το θε... ως προς τα ερωτήματα που με ρωτήσατε, ως προς το TTIP, στον κύριο Ως προς το θέμα της συνεργασίας Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου σε θέματα προτύπων, τόνισα την, από την πρώτη στιγμή την πρόθεση της ελληνικής προεδρίας να εργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο πιο συστηματικά μπορούμε για την επίτευξη κοινού, κοινών αποφάσεων. Ως προς το θέμα της ε, TTIP ε, και τα... αναφορικά με την πρόοδο της διμερείς συμφωνίας ως προς το θέμα της ΣΕΤΑ γνωρίζουμε ότι έχει επιτευχθεί η συμφωνία επί της πολιτικής αρχής αλλά ακόμα γίνεται συζήτηση για την ειρωστικοποίηση ε, των τελικών κειμένων και υπάρχει επικοινωνία και μεταξύ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως αντιλαμβάνομαι, ω προ την προσπάθεια ολοκλήρωση αυτών των κειμένων. Δεν έχουμε λάβει επίσημα τελικά κείμενα, όπω δεν έχετε λάβει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό άρα πρέπει να δούμε κατά πόσο θα υπάρξει τελικά πρόοδος επικειμένων στη διάρκεια της Προεδρίας. Όσο στο TTIP θα προσπαθήσουμε, εκμεταλλευόμενοι και το άτυπο Συμβούλιο της Αθήνας, να προχωρήσουμε τις συζητήσεις μετά την ε, συνάντηση που θα έχει πραγματοποιηθεί μεταξύ της Επιτροπής και του Αμερικανού διαπραγματευτή στις 17 ε, Φεβρουαρίου. Οι σχέσεις καλής γειτονίας το θέμα της, των εμπορικών συμφωνιών θεωρούμε ότι συμβάλλει στη σταθερότητα της περιοχής. Και η Ευρώπη αντιμετώπισε θέματα τα τελευταία χρόνια και θέματα παραδείγματο χάρη λαθρέα μετανάστευση, τα οποία ήταν αποτέλεσμα πολιτικών και οικονομικών προβλημάτων που στην ευρύτερη γειτονιά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούμε λοιπόν ότι η προώθηση εμπορικών συμφωνιών και γι' αυτό τέθηκε και ω προτεραιότητα τη ελληνική προεδρία με τι χώρε του Μεσογείου, όπου υπάρχει ήδη ένας ανοιχτός διάλογος, θα συμβάλλει σε αυτή την ε, κατεύθυνση. Ως προς το θέμα της Κίνας, υπήρχε και το Συμβούλιο έλαβε σοβαρά υπόψη τότε όταν δώσαμε τον Οκτώβριο τη διαπραγματευτική εντολή τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει πρόσβαση ε, στις αγορές της Κίνας και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα το οποίο παραμένει στην πρώτη γραμμή των διαπραγματεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως προς το θέμα των σχέσεων με την ε, Ανατολική Ευρώπη και τη Ρωσία είναι λίγο θέματα τα οποία ξεφεύγουν και της δικιάς μου άμεσης αρμοδιότητας κάποια από αυτά ε, ως προς το θέμα του εξωτερικού εμπορίου και έχουν να κάνουν με τη γενικότερη έκφραση της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, το Συμβούλιο Εξωτερικού Εμπορίου είχε, είχε από την πρώτη στιγμή στηρίξει τις, ε, του East ε, Europe Neighborhood και παραμένουμε σε αυτή τη γραμμή. Σας θυμίζω ότι για το θέμα της Ουκρανίας πριν την ε, αποτυχία της διαπραγμάτευσης η Ευρώπη είχε θέσει και κάποια πολιτικά benchmarks τα οποία εξακολουθούν να αντανακλούν και την άποψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε θέματα εμπορίου. Κύριε Δεύτερος ερωτήσεων. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον Υπουργό για την παρουσίασή του. Ένα άλλο θέμα. Δεν ανέφερε νομίζω ο Υπουργός καθόλου την Ινδία Αυτό σημαίνει ότι η προόδος με την Ινδία είναι πολύ αργή ή για ποιο λόγο, ο πάση δεν αναφέρθηκε η Ινδία καθόλου. Μετά, για τη ΣΥΤΑ και την, το Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών των Επενδυτών. Ε, εδώ υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον της ελληνικής κοινωνίας στα θέματα αυτά δεδομένο, δεδομένης της ιστορίας με τα ορυχεία χρυσού στη Βόρεια Ελλάδα, το Ελντοράντο και τα λοιπά, εκεί η ελληνική κοινωνία ε, αντέδρασε. Ε, αν η κυβέρνηση ή μια μελλοντική, κυβέρνηση αποφάσισε ότι τα δικαιώματα του περιβάλλοντος προέχουν ε, τότε ε, θα δημιουργηθεί πρόβλημα με την ε, συμφωνία οπότε είναι σημαντικός ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Άλλο ερώτημα για τη Μεσόγειο. Θα γίνει τον Ιούνιο νομίζω ότι έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο η συνάντηση διάσκεψη για τη Μεσόγειο θα γίνει αλλά αναβλήθηκε θα γίνει διάσκεψη αυτή για να υπάρξουν πιο βαθιές και πιο στενές σχέσεις με τις χώρες της ε, λεκάνης της Μεσογείου γιατί και αυτές θα βοηθήσουν στην ανάπτυξη τέλος μπορεί να το είπατε αλλά δεν το πήρα είδηση ε, έχετε ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα ε, για, τις, ε, για τη σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Θα τελειώσουμε φέτος. Εγώ έχω τρεις ανησυχίες και θα ήθελα να σας τις παρουσιάσω κύριε Υπουργέ και να ακούσω και την θέση σας, την άποψή σας. Πρώτον, όσον αφορά τις ε, θέσεις κάποιων κρατών μελών, την ε, αντίθεση κάποιων κρατών μελών όσον αφορά τις εμπορικές πολιτικές και σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είδαμε παραδείγματος χάρη ότι σε πολλές ε, χώρες υπάρχει αντιπαράθεση, στη Γαλλία, δεν ξέρω και στη χώρα σας, κατά του εμπορίου, κατά των εμπορικών συναλλαγών. Βλέπουμε να υπάρχει μία αντίθεση και βεβαίως το θέμα των ε, ισορροπημένων εμπορικών σχέσεων, των συμμαχιών. Αυτό είναι ένα θέμα που εξελίσσεται, που αλλάζει. Πώς ε, αντιμετωπίζει το Συμβούλιο το θέμα αυτό. Πώς βλέπετε το θέμα αυτό εσείς. Βλέπετε κάποιο κίνημα, κάποια κίνηση. Θεωρείτε ότι το να έρχεται κανείς από μια χώρα με κρίση, με παρουσία τρόικας, με τρομερή κοινωνική κρίση, σας κάνει να είστε πιο κοντά στο πρόβλημα ή πιο κοντά στη λύση. ο ρόλος του εμπορίου όσον αφορά την οικονομική ανάπτυξη, όσον αφορά την μελλοντική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος θα μπορούσε να είναι. Βεβαίως και εδώ χρειαζόμαστε πολιτική συζήτηση, δεσμεύσεις. Ποια είναι η θέση του Συμβουλίου, τι θέλει να κάνει το Συμβούλιο ή τι κάνει το Συμβούλιο. Δεύτερον, εγώ είμαι εισηγητής και διαπίστωσα ότι εδώ υπάρχει ουσιαστικά για το θέμα του TTIP, για την προστασία των δεδομένων, για το θέμα της επίληψης των διαφορών ε, σε θέματα επενδύσεων, Υπάρχουν πολλά εκκρεμή θέματα και επειδή έχω ιδιαίτερο ενδιαφέρον σαν εισηγητής για το θέμα αυτό, θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς βλέπετε εσείς αυτήν την αυξανόμενη αντίθεση για το θέμα αυτό. Τι θα κάνουμε εμείς σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, σαν Συμβούλιο, θα περιμένουμε όπως έγινε και με την Άκτα, γιατί όσον αφορά το θέμα της Άκτα, κάποια από αυτά τα θέματα είχαν προκύψει και βεβαίως επειδή υπήρξε μια οργανωμένη αντίθεση και αντίδραση κατά της άκτα, τα θέματα αυτά παρέμειναν και εμείς καταφέραμε τελικά να σκοτώσουμε το άκτα. Τι θα κάνει το Συμβούλιο τώρα. Τι θα κάνει το Συμβούλιο έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα λανθασμένα επιχειρήματα τα εσφαλμένα επιχειρήματα και όλα αυτά τα κινήματα κατά του εμπορίου. Γιατί εγώ πραγματικά όταν ακούω ότι στη Γαλλία οι περισσότεροι είναι κατά αυτών των ε, συμφωνιών για το εμπόριο. Και αυτά τα επιχειρήματα δεν είναι σωστά, δεν ευσταθούν. Αν ρωτήσετε όμως, αν κάνετε μια δημοσκόπηση στη Γαλλία, για τα θέματα παραδείγματο χάρη της ε, ορμόνης στο κρέα. παραδείγματο χάρη θα δείτε ότι υπάρχει πάρα πολύ έντονη αντίδραση και ότι υπάρχουν πάρα πολλά αβάσιμα επιχειρήματα. Τρίτη ανησυχία την οποία θα ήθελα να σας ε, παρουσιάσω είναι Υπάρχουν ακόμα τρία ή τέσσερα εκρεμή θέματα νομοθετικού περιεχομένου. Σήμερα η ελληνική προεδρία δεν έχει έξι μήνες, αλλά τέσσερις λόγω των εκλογών. Και βεβαίως υπάρχουν ουσιαστικά θέματα, τα οποία είναι εν εξελίξη. Για μένα το πιο σημαντικό είναι η νομοθεσία όσον αφορά την εφαρμογή και βεβαίως το TDI θεωρώ ότι δεν είναι ρεαλιστικό να θεωρήσει κανείς ότι όλα αυτά θα ολοκληρωθούν. Αλλά όσον αφορά τις ε, ρυθμίσεις για την εφαρμογή όσον αφορά τον εφαρμοστικό κανονισμό αλλά και όσον αφορά τις αποζημιώσεις και τις πληρωμές, θα ήθελα να ξέρω πώς ε, εσείς βλέπετε την διεκπαιρέωση αυτών των δύο θεμάτων, καθότι έχετε δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίξει εδώ το ρόλο της ε, όσον αφορά το γεφύρωμα του χάσματος, καταρχήν μεταξύ των ε, διαφορετικών θέσεων. Εμείς, εμείς σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαστε διατεθειμένοι να βρούμε μια συμβιβαστική λύση. Βεβαίως εδώ περιμένουμε και επισκηνήσεις από μέρους Συμβουλίου. Πρόκειται για ένα πακέτο μέτρων. Και δεν είμαι σίγουρος ότι το Βουλίο πρόκειται να συμφωνήσει με αυτή την προσέγγιση. Περιμένουν περαιτέρω υποχωρήσεις ε, από μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Από ό,τι ξέρω, δεν είναι ε, δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει άλλες υποχωρήσεις ε, στα θέματα αυτά. Και βεβαίως το non-paper της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρέπει οπωσδήποτε, αυτό είναι προϋπόθεση, να γίνει δεκτό. Τι θα κάνει το Συμβούλιο. Δεν μπορεί το Συμβούλιο να τα θέλει όλα δικά του. Δάμε ένα συμβιβασμό. Πρόκειται για ένα σύστημα με δύο νομοθετικές αρχές και δεν είναι δυνατόν τον Συμβούλιο να θέλει και για τα δύο αυτά θέματα, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο, να περάσουν όλες οι δικές του θέσεις. Τις επόμενες δύο εβδομάδες λοιπόν θα πρέπει να επιτύχουμε αυτήν την, αυτόν τον συμβιβασμό, αλλιώς θα υπάρξει πλήρης αποτυχία, δηλαδή δεν θα υπάρξει νομοθεσία. Και αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι η Προεδρία τι προτίθεται να κάνει. Μπορεί να πιέσει το Συμβούλιο, να τους πείσει ότι πρέπει και οι δύο να κάνουν κάποιες υποχωρήσεις για να υπάρξει αυτή η νομοθετική πρόταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έκανε αρκετές υποχωρήσεις. Και είμαστε διατεθειμένοι πραγματικά να υποχωρήσουμε και σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Εάν όμως το Συμβούλιο είναι διατεθειμένο να υποχωρήσει όσον αφορά τις αδικαιολόγητες αυτές απαιτήσει για την επιτροπολογία. Αυτό είναι ένα πολύ ισχυρό μήνυμα που θα θέλαμε να το περάσετε στο Συμβούλιο. Το θέμα της επιτροπολογίας δεν μπορεί εδώ να καλύψει όλα αυτά τα θέματα. Και νομίζω ότι οι συνάδελφοι στο Συμβούλιο δεν το έχουν διαπιστώσει, δεν το έχουν κατανοήσει αυτό. Δεν πρόκειται να επιτρέψουμε κατάχρηση της αρχής της επιτροπολογίας Και πραγματικά εδώ θα παραμείνουμε σε αυτό που προβλέπει η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Και δεν υπάρχει εδώ καμία απολύτως δυνατότητα εξαίρεσης ε, για το Συμβούλιο. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει η Ελληνική Προεδρία εδώ να πετύχει. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. I'll Θα προσπαθήσω να απαντήσω με λιγότερο εύγλωτο, αλλά με τον ίδιο, με παρόμοιο τρόπο. Να απαντήσω στις ερωτήσεις ε, με τη σειρά που τέθηκαν. Για την Ινδία. Βεβαίως και θεωρούμε σημαντική και στη σχέση μας με την Ινδία, αλλά ως Προεδρία στο λίγο χρόνο που έχουμε πρέπει να κάνουμε επιλογές και να θέσουμε προτεραιότητες για συμφωνίες που είναι είτε πιο όριμες είτε έχουν μεγαλύτερη ε, πιθανότητα υλοποίησης. Και παρουσιάσαμε σε σαφή τρόπο τις χώρες στις οποίες ε, θα δώσουμε έμφαση για την Προεδρία μας για τις ε, επενδύσεις που αναφέρεται στις, στους φυσικούς πόρους στη Βόρεια Ελλάδα. Βεβαίως η Ελλάδα όπως κάθε χώρα της Ένωσης θέλει να προσελκύσει επενδύσεις και νομίζουμε ότι οι επενδύσεις δημιουργούν θέσεις εργασίας και μείωση της φτώχειας, λαμβάνοντας ε, η χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων είναι σημαντική και για την Ευρώπη, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και για ασφάλεια στον τομέα της ενέργειας. Η ειδική επένδυση που αναφέρεται στη Βόρεια Ελλάδα σέβεται βεβαίως ε, τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές και πήρε άδεια. Οποιαδήποτε προσπάθεια να, να αλλάξει, να σταματήσει την επένδυση απέτυχε και τα επεισόδια βίας ε, ομάδων ε, κατά των αρχών της χώρας διώχθηκαν όπως θα συμβαίνει σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα. Δεν προβλέπουμε... Καταλαβαίνω τι εννοείται. Εγώ σας λέω ότι υπήρξε βία οι υπάλληλοι των εταιριών ε, υπέστησαν νύχτα επίθεση, ε, τους ε, έριξαν βενζίνη, καταστράφηκαν προϊόντα και δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς που δεν θέλει να καταδικάσει μια τέτοια πράξη βίας και στο κοινοβούλιο εδώ και αλλού. Σε ό,τι αφορά, όπως είπα μάλλον, οι επενδύσεις δουλεύουν και οποιαδήποτε ρήτρα ε, διαιτησία δεν επηρεάζει την ελληνική δημοκρατία. Εμείς πιστεύουμε στο κράτο δικαίου και επιτρέπουμε στου επενδυτέ να έχουν ε, το δικαίωμα πρόσβαση στα δικαστήρια, στη δικαιοσύνη. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα για τις ΗΠΑ, εμεί το εξάμεινό μα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επέλθει πρόοδο στο TTIP. Όταν ε, κάνουμε την ανασκόπηση το Φεβρουαρίου θα δούμε αν το χρονοδιάγραμμα είναι αισιόδοξο ή απεσιόδοξο, όχι τώρα. Ευχαριστώ πρόεδρε που πήρατε το λόγο και θέσατε πιο πολιτικές ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω να κρατήσω μια ισορροπία μεταξύ Εθνικού Υπουργού και Προεδρεύοντος του Συμβουλίου. Δύσκολη ισορροπία, ιδίω όταν θέλετε μια σειρά θεμάτων με εθνική διάσταση είναι σαφές σε πολλά κρατημέλη ότι, πολλά, ότι οι πολίτες θέτουν πολλά ερωτήματα. Η πρόσφατη οικονομική κρίση που επηρεάζει βαθιά, πολύ βαθιά πολλές ευρωπαϊκές χώρες και οδήγησε σε ύφεση ολόκληρη την Ευρωζώνη είναι κάτι που οι πολίτες ζητήσουν εν ώψη των ευρωεκλογών και ως πολιτικοί θα πρέπει να παρουσιάσουμε λύσεις κατά την άποψή μας. Το εμπόριο κατά την άποψή μας είναι κομμάτι της λύσεις. Η ανάκαψη της ελληνικής οικονομίας που ξεκίνησε και έχει δημιουργήσει και πρωτογενές πλεόνασμα και εμπορικό πλεόνασμα έγινε διότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές και αγαθών και υπηρεσιών που απετέλεσαν βασική κατευθυντήρια γραμμή για να έχουμε για πρώτη φορά ε, για το, δεύτερο, για το 2014 αναθεώρηση προς τα άνω του πλεονάσματος. Αυτό ισχύει και για ολόκληρη την Ευρώπη. Το εμπόριο δημιουργεί θέσεις εργασίας και έχει πλεονεκτήματα για όλους μας. Γι' αυτό συζητούμε και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και Επιτροπής όλες αυτές τις εμπορικές συμφωνίες. Η Ευρώπη πρέπει να απαντήσει στους πολίτες λέγοντας ότι αυτό που κάνουμε πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και ο στόχος είναι η μείωση της φτώχειας και της ανεργίας. Για το TTIP τώρα το Φεβρουάριο θα ανοίξουμε το Συμβούλιο σε άτομα που θα έρθουν από τον κλάδο της βιομηχανίας για να συζητήσουμε για το θέμα του TIP, περνώντα και ένα μήνυμα προς το κοινό, ε, τονίζοντας δηλαδή τα πλεονεκτήματα που θα έχει η TTIP για την ευρωπαϊκή οικονομία. Βεβαίως ε, υπάρχει ένας ε, κίνδυνος να μπλοκάρουμε κάπου, πάντα υπάρχουν σημεία που πρέπει να είμαστε προσεκτικοί είναι σημαντικό για όλους μας να μπορούμε να περνάμε καλύτερα επικοινωνιακά τα πλεονεκτήματα της συμφωνίας αυτής. Μα ένα από τα θέματα μου συζητείται. ISTS. Ποια άποψη έχει το Συμβούλιο για το αν το ISPS θα πρέπει να είναι στο TDIP ή όχι. Με αυτό θα συζητήσουμε το Φεβράριο στο Συμβουλίο είναι πολύ κρίσιμο θέμα. Σωστά το θέσατε. επίση, καταλαβαίνω ότι και η Επιτροπή έστειλε επιστολή στην Επιτροπή σα στο Συμβούλιο με μια σειρά θεμάτων για το ISDN, ISDS 4TT, για το TTIP. Το θέμα των νομοθετικών φακέλων προφανώς χρειάζεται να ασκήσουμε πίεση στους συναδέλφους μας για να μπορέσουν να προχωρήσουν ταχύτερα τα ντοσιέ καταλαβαίνουμε στον τομέα της χρηματοοικονομικής ευθύνης υπάρχει ένα κείμενο συμβαστικό από την Επιτροπή που έγινε δεκτό από εσά ως πακέτο. Θα συζητηθεί το θέμα στις 29 Ιανουαρίου ε, στο Συμβούλιο για να δούμε ποια είναι η άποψη των κρατών Εμείς θα καταβάλουμε προσπάθεια για να βρεθεί συμφωνία στα πλαίσια αυτά. Σε ό,τι αφορά Τώρα, σε ό,τι αφορά τον, ε, εκτελεστικό, τον εφαρμοστικό κανονισμό, σήμερα θα βγει ένα κείμενο της Προεδρίας με τις απόψεις μας για το θέμα. Καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει πολύ περιορισμένος χρόνος στη διάθεσή μας για να βρεθεί λύση μέχρι το Φεβρουάριο. Θα είναι μια μεγάλη επιτυχία και για τις δύο πλευρές αν πετύχουμε Αν, αντί λοιπόν να λέμε ότι θα ήταν αποτυχία αν δεν το κάναμε, ας πούμε να πούμε ότι είναι επιτυχία αν το κάνουμε. Αισιοδοξία. Μπράβο, χαίρομαι. Κάποιος άλλος. Ε, ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να ξαναμιλήσω. Δυστυχώς λείπουν πολλοί συνάδελφοι. Έχω και μια σειρά ε, συμπληρωματικών ερωτήσεων. για το TTIP. Σωστά είπατε ότι πρέπει να έχουμε επίγνωση της προσοχής που θα δοθεί από το κοινό, αλλά τις επιχειρήσεις και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Γι' αυτό ρωτώ, στο τέλος του μήνα η Επιτροπή θα θεσπίσει μια επιτροπή διαβούλευσης που θα συνοδεύει την περαιτέρω δουλειά της διαπραγματευτικής ομάδας. Πώς εμπλέκεται το Συμβούλιο σε αυτό. Θα υποστηρίζετε την θέση του Κοινοβουλίου να υπάρξει μόνιμη σύνδεση μεταξύ των συνομοθετών για να καταλάβουμε πώς και ο Δήμος, το κοινό παρακολουθεί τις διαπραγματεύσεις. Επίσης είπατε ότι θα καλέσετε στο δεύτερο γύρο κοινό. Θα σας έλεγα να καλέσετε και άλλες ομάδες, συνδικάτα, περιβαλλοντικές οργανώσεις που ανησυχούν για θέματα TTIP. Οι ανησυχίε τους πρέπει να αντιμετωπιστούν και να απαντηθούν με όσο περισσότερη διαφάνεια γίνεται. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να περάσετε στο κοινό ότι εδώ δεν παίζει μόνο το θέμα του εμπορίου και του ωφέλους των επιχειρήσεων αλλά και του ωφέλους του κοινού, των πολιτών. το οποίο είναι σημαντικό για όλους και τις 28 χώρες αλλά και για το ελληνικό κοινό. Ο καθηγητής κ. Μορέρια περιέγραψε τις προσδοκίες που υπάρχουν από την Προεδρία σας. Πριν τις ευρωεκλογέ πρέπει να μπορέσουμε να περάσουμε στους πολίτες ότι αυτή η Ένωση κάνει κάτι καλό για τον κόσμο. Μια ακόμα ερώτηση. Είπατε να είσαστε σύντομοι ποια είναι τα κανονιστικά στάνταρ που θέλετε να διαπραγματευτείτε με τις ΙΠΑ για να απαντήσετε στις προσδοκίες. Ποια είναι τα στάνταρ σε περιβαλλοντικό και εργασιακό επίπεδο. Η διαπραγμάτευση γίνεται από την Επιτροπή, όχι από το Συμβούλιο. Κύριος Καζάκ. Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος. Ακούσαμε τον Υπουργό να αναφέρει τη σημασία αυτών των εμπορικών διαπραγματεύσεων και το κατά πόσο χρειάζεται η μέγιστη προστασία που μπορεί να επιτευχθεί. Εγώ κατάλαβα ότι κατά τη διάρκεια των συναντήσεων που είχαμε με τους Έλληνες εκπροσώπους του Κοινοβουλίου που αναφερόταν σε ελληνικά προϊόντα όπως η φέτα, οι ελιές καλαμάτας ήταν πάρα πολύ σημαντικές και αυτό βεβαίως ισχύει και για άλλες χώρες που έχουν παρόμοια προϊόντα τα οποία χρήζουν προστασίας στις τρίτες αγορές κυρίως. Πιστεύετε λοιπόν ότι κατά τη διάρκεια αυτών των πολύ σημαντικών διαπραγματεύσεων με τις ε, Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και με άλλους εμπορικούς μας εταίρους, οι προσδοκίες των ε, καταναλωτών όσον αφορά αυτές τις ονομασίες προέλευσης, αυτά τα προϊόντα, τα πολύ συγκεκριμένα, θα στεφθούν με επιτυχία, γιατί ξέρουμε ότι σε πολλές άλλες ε, χώρες δεν υπάρχει τέτοιου είδους παράδοση. Θα μπορέσει να είναι πιστική εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή. Um, Αναφερθήκατε και στην ε, φέτα. Καταλαβαίνω ότι η πρώτη ερώτηση του Χέλμουτ Σόλτς δεν ήταν τόσο σαφής. Έχω την εντύπωση ότι περίμενα να ακούσει κάτι για την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και για το κατά πόσο θα μπορούσαν να συμμετάχουν εκεί και εκπρόσωποι των μη κυβερνητικών οργανισμών και άλλων ενώσεων. Η συμμετοχή και άλλων παραδείγματος χάρη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις θα μπορούσε να ληφθεί υπόψη. Είναι πολύ σημαντικό το να εισακουστούν οι απόψεις όχι μόνο της, των επιχειρηματιών και των εταιριών αλλά και άλλων ομάδων ε, που ασχολούνται με την προστασία των περιβάλλοντων κτλ. Όντως χρειάζεται να είναι μεγάλο το εύρος των συνομιλητών μας και η Κομισιόν αν κατάλαβα καλά θα κάνει κάτι τέτοιο. Η Κομισιόν προωθεί ένα ευρύ διαπραγματευτικό, διαβουλευτικό πλαίσιο για αυτό το θέμα. Αλλά αυτό είναι πρωτοβουλία της Κομισιόν, δεν είναι του Συμβουλίου. Ε, για την, όσον αφορά την Αθήνα θα κάνουμε... Ε, μια σχετική, μια κάποια διάσκεψη αν θέλετε αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε διαβουλεύσεις στο εύρος που θα τις κάνει η Κομισιόν αλλά βεβαίως θα σας ενημερώσουμε σχετικά τώρα ε, για την άλλη σας ερώτηση οι παραδόσεις των διαφόρων χωρών είναι διαφορετικές στην περίπτωση του Καναδά ας πούμε είδαμε τι γίνεται αλλά κατά την άποψή μας ε, η ονομασία προέλευσης οι ενδείξει για δεν είναι ε, προστασία και εκεί τελειώνει. Είπα και αν επιληθεί το πρόβλημα, αν θέλετε, μέσω γεωγραφικών ενδείξεων, λύνεται με όλα τα προβλήματα ε, επιλύονται. Όχι, υπάρχει και θέμα τιμών και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα για τις γεωγραφικές ενδείξεις, βέβαια, μέσα στα πλαίσια του της συμφωνίας TTIP ε, έχετε δίκιο ε, είναι, παίζουν μεγάλο ρόλο εκεί στην τελική εκδοχή σίγουρα θα υπάρχει μεγάλη επαρκής προστασία των ευρωπαϊκών γεωγραφικών ενδείξεων. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ για όλη τη συζήτηση που έγινε εδώ. Χαιρόμαστε που είσαστε εδώ κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Προχωράμε, σημείο 5. Νομοθετικός φάκελος. Νομοθετικό κείμενο δηλαδή. Προσαρμογή των κοινοτικών στατιστικών εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες στον ε, νέο κανονισμό για την λεγόμενη επιτροπολογία και την ανάπτυξη κατεξουσιοδότηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. Είμαι εισηγητής. Οι τροπολογίες περισσότερες από μένα κατατέθηκαν. Υπάρχουν και κάποιες που έχει υποβάλει ο κύριος Οντί που πρέπει να σας πω θα μπορούσα να τις και εγώ και συμφωνώ λοιπόν με τις τροπολογίες του αδελφού Οντί που έχουν στόχο να υπάρξει υποχρεωτική προθεσμία για την ενοποίηση του κανονισμού μετά την τροποποίηση του κανονισμού. Για τις δικές μου τροπολογίες τώρα, ήταν μια μορφή επιτροπολογίας ε, που e που ήταν Regulated Procedure with Scrutiny. περίεργη διαδικασία ήδη τότε. Η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, αυτό το αφορούσε την κανονιστική το να χορηγηθεί στην Επιτροπή μια μορφή κανονιστικής αρμοδιότητας. Δηλαδή δίναμε στην Επιτροπή πριν τη Λισαβόνα με ένα είδος εξουσιοδότησης. Οι νομικές πράξεις λοιπόν που είχαν εκχωρηθεί σε εισαγωγικά στην Επιτροπή ήταν ε, κανονιστικού χαρακτήρα, είχαν κανόνες. Και με έκπληξη είδα ότι η Επιτροπή αντί να αλλάζει όλες ε, τις εφαρμοστικές πράξεις, ε, τις εκτελεστικές πράξεις σε κατεξοδότηση πράξης έκανε κάποια επιλογή. Κάποιες εκτελεστικές τις έκανε κατεξοδότηση και κάποιες τις κράτησε ως εκτελεστικές χωρίς παρέμβαση δηλαδή του Κοινοβουλίου, διότι όπως ξέρετε οι εκτελεστικές πράξεις αποφασίζονται από την Επιτροπή και ελέγχονται από το Συμβούλιο, τα κράτη-μέλη, όχι από το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και αυστηροί όταν έχουμε να εξετάζουμε ποιο είναι το σύνολο μεταξύ εκτελεστικών και, εκτελεστικών και κατεξουσιοδότηση πράξου, γιατί ανήκουν σε τελείω διαφορετικές οικογένειες. Αποφάσισα λοιπόν και εγώ να αλλάξω τα πάντα και να τα κάνω κατεξουσιοδότηση πράξη, διότι κατά άποψή μου όλε όλες οι πράξει ε, που περιλαμβάνονται εκεί περιλαμβάνουν κανόνε ρυθμίσει και σε μια κοινοβουλευτική δημοκρατία θα πρέπει να τροποποιούνται βάσει του από το Κοινοβούλιο και όχι να ασκούνται από το εκτελεστικό όργανο χωρίς εξουδότηση από τον νομοθέτη. Γι' αυτό αποφάσισα να καταργήσω ό,τι έχει να κάνει με την επιτροπολογία, να διαγράψω ό,τι έχει να κάνει με τις εκτελεστικές πράξεις και να τις κάνω όλες κάτι εξουσιοδότηση. Αυτός είναι ο στόχος των τροπολογιών μου. Περιμένω τα σχόλιά σας. Δεν βλέπω κάποιον άλλον. Άρα βλέπω ότι μάλλον υπάρχει συνένεση. Κομισιόν. Η κυρία Φιγκέιρα. Έλενα. Παρακαλώ. Muito Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν να σας πω ότι το σχέδιο έκθεσης και η τροπολογία σας καταρχήν αντιμετωπίζονται με θετικό τρόπο από την Επιτροπή. Μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πιστεύω ότι υπάρχει συνάφεια και θα μπορέσουμε στην πρώτη ανάγνωση να προχωρήσουμε. Καταρχήν όσον αφορά τη συλλογή στοιχείων για την εμπορική πολιτική, ιδιαίτερα σε τρίτες χώρες και δεύτερον όσον αφορά το θέμα της επιτροπολογίας και της μεταφοράς μέσω του συστήματος ESSE e, που Εξάλλου δημιουργήθηκε, ιδρύθηκε για αυτόν τον σκοπό το 2009 με το άρθρο 299. Ουσιαστικά λοιπόν εδώ παρακολουθείτε και ακολουθείτε η λογική αυτής της θεσμικής ε, συμφωνίας, ιδιαίτερα για τις ε, κατεξουσιοδότηση πράξεις. Η Επιτροπή λοιπόν μπορεί να θεωρήσει ότι όσον αφορά τον περιορισμό σε χρόνο που προτείνει η αντίστοιχη τροπολογία μπορεί να γίνει δεκτή. Παρόλα αυτά η Επιτροπή δεν μπορεί να στηρίξει την χρήση των κατεξουσιοδότηση πράξεων για μέτρα που αφορούν την κωδικοποίηση, την τεχνική κωδικοποίηση των στατιστικών δεδομένων. Θα ήθελα εδώ να υπογραμμίσω το γεγονός ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής όσον αφορά τα νομικά εργαλεία που έχουν επιλεγεί βασίζεται σε μια εις ανάλυση όλων των θεμάτων. Και τέλος, και αυτή είναι ίσως και η πιο σημαντική μου παρατήρηση, ανησυχούμε όσον αφορά τις τροπολογίες που αμφισβητούν το δεύτερο σκοπό της πρότασής μας και η στρατηγική για μια νέα ε, δημιουργία ενός στατιστικού συστήματος, βάση δηλαδή της πρωτός του 2009, και αυτό βεβαίως αναφέρομαι εδώ σε όλες τις δραστηριότητες που καλύπτουν ε, την ε, ευρωπαϊκή στατιστική σε όλους τους τομείς και βεβαίως εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μπορεί να ασκήσει την ε, δυνατότητα άσκηση αυτής της στατιστικής πολιτικής σε όλους, σε όλους υπογραμμιζώ τους τομείς. Προτείνεται λοιπόν να σβηστεί η αναφορά στο SSE, κάτι που δεν μπορεί να δεχτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θεωρούμε λοιπόν ότι εδώ θα πρέπει να ξαναεξετάσετε αυτές τις ε, τροπολογίες. Πρόεδρος, εγώ δεν αναφέρομαι εδώ στην επιτροπολογία, επαναλαμβάνω, αλλά αμφισβητώ σε αυτές τις περιπτώσεις της κατεξουσιοδότηση πράξης. Ζητάει κάποιος το λόγο, δεν βλέπω κανέναν. Uh, Βλέπω εδώ ότι το Συμβούλιο δεν θα λάβει στο άμεσο μέλλον θέση για το θέμα αυτό, άρα δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία. Θα δούμε τι θα γίνει στην Ολομέλεια. Άρα δεν μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία πρώτης ανάγνωσης. Αύριο εμείς θα ψηφίσουμε. Και το Μάρτιο στην Ολομέλεια βεβαίως. Και περνάμε στο σημείο 6. This is an oral question. Πρόκειται για μια προφορική ερώτηση που αφορά ουσιαστικά τα αντιδοτικά μέτρα της λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας κατά του ίνου που εισάγεται στην Κίνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για μια πολιτική απόφαση που βεβαίως είναι μια αντίδραση της Κίνας για την ευρωπαϊκή απόφαση όσον αφορά τα ηλιακά πάνελ. Πρόκειται για μέτρα anti-dumping και βεβαίως ε, εδώ βασιζόμαστε και σε διαπραγματεύσεις που γίνονται στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Ακούσαμε την ε, Επιτροπή το Δεκέμβριο. Ποιος θα ήθελε να πάρει το λόγο για το θέμα αυτό. Ο κύριος Σόλτ. Thank you, Mr. Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είστε ο εισηγητής για την Κίνα. Ναι. Καταρχήν, ποια είναι η ουσία όλης αυτής της αντιπαράθεσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακολουθήσουμε αυτή την κατεύθυνση. Και το τελευταίο σημείο είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε. Δηλαδή, προσπαθούμε εδώ να ευαισθητοποιήσουμε όσον αφορά την πολιτική προσέγγιση. Είναι ένα εμπορικό θέμα, ναι. Αλλά προσπαθούμε να βρούμε μια λύση γενικότερη και θα ήθελα πραγματικά να ακούσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κατά πόσο υπάρχει η περίπτωση να βρεθεί λύση. Ο κύριος Κορέα από το ΕΛΚ. Η κυρία Κορέα, συγγνώμη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, τον, Ιανουάριο, τον Ιούνιο του 2013 ξεκίνησε διαδικασία αντιτάμενη από την Κίνα στις εισαγωγές ε, ίνου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων από, αυτών αποτελεί επίθεση από πλευράς ε, Κίνας στην απόφαση που έλαβε στις 5 Ιουνίου η Επιτροπή να επιβάλλει προληπτικά μέτρα αντι-dumping παρότι στις 27 Ιουλίου αναγγέλθηκε ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ Ένωσης και Κίνας για, ε, για τα πάνελ που Κίνας, η συμφωνία αυτή δεν ε, οδήγησε στην πάυση της διαδικασία ε, έρευνας που έχει ξεκινήσει για τις εισαγωγές ευρωπαϊκού κρασιού στην Κίνα. Θέλω να υπογραμμίσω σήμερα ότι ο Ευρωπαϊκός Ίνος είναι 65% των εισαγωγών κρασιού στην συνολικά. Η κατάσταση αυτή ανησυχεί ιδιαίτερα τον αμπελοϊνικό τομέα της Ευρώπης, ιδίως τις τρεις κύριες χώρες εξαγωγής, Ισπανία, Ιταλία και Γαλλία, καθότι το περιθώριο πέραν του ότι έχει οικονομικό κόστος για τον αμπελοϊνικό τομέα της Ένωσης, επηρεάζει αρνητικά την καλή φήμη του... μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά διότι η διερμηνία δεν προλαβαίνει. Ναι, ναι, έλεγα ότι αυτό επηρεάζει αρνητικά την ε, καλή φήμη του κλάδου σε διαδικασίες όπου κατηγορείται ότι προβαίνει σε παράνομες εμπορικές πρακτικές. Για το λόγο αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό το Κοινοβούλιο να έχει την ευκαιρία να απαιτήσει, να ζητήσει, να εξετάσει τον Επίτροπο Εμπορίου για θέματα που ανησυχούν ιδιαίτερα τον ε, αμπελονικό κλάδο στην Ένωση, ιδίως δε την υφιστάμενη κατάσταση των διαπραγματεύσεων κλάδο για να υπάρξει μια φιλική λύση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε διακοπή της ε, διαδικασίας παραπομπής ε, χωρίς να, υπάρξουν, χωρίς να είναι επιβλαβής για, τον, ε, για το κρασί στην Ένωση και χωρίς να υπάρχουν άλλες, ε, άλλα αντιμπορικά αντίμετρα από πλευράς Ένωσης ή από πλευράς άλλων χωρών ε, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα μέτρα προστασίας, εμπορικής προστασίας. ΕΛΚ, κυρία Μαρία, Ευχαριστώ πρόεδρε. Να συγχαρώ του συναδέλφου ε, της ΣΥΝΤΑ για την προφορική ερώτηση προ την Επιτροπή. Η Επιτροπή Γεωργίας ε, θεωρεί πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Το ξεκίνημα δηλαδή, από τότε που ξεκίνησαν οι δυσκολίε με την Κίνα και εγώ ως ε, ε βουλευτής είχα θέσει γραπτές ερωτήσει προς την Επιτροπή για να ζητήσω τι μέτρα λαμβάνει η Επιτροπή και η Επιτροπή πάντα απαντούσε εγγράφους ότι ξεκινούν διαπραγματεύσεις προσπαθώντας να λύσουν το πρόβλημα. Γνωρίζουμε ωστόσο ότι οι παραγωγή ίνου στην Ευρώπη συνεχίζουν να παραπονούνται ότι δεν λύνεται το πρόβλημα. Ξέρετε ότι η Επιτροπή Γεωργίας ξεκίνησε ε, να εξετάζει την έκθεση για την προώθηση των ε, γεωργικών προϊόντων που είμαι εισηγήτρια. Ο κ. Τσόλος τονίζει, ο Επίτροπος, ότι τα κονδύλια που θέλει να δώσει, της, να δώσει Ένωση για την προώθηση του, των προϊόντων είναι για τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων ε, χώρες της, ε, της Ανατολικής Ασίας. Για το λόγο αυτό η ερώτηση είναι εξαιρετικά επίκαιρη. Θα διαδώσουμε 200 εκατομμύρια ευρώ, 200 εκατομμύρια ευρώ για δράσεις προώθησης και ο στόχος που θέτουμε ε, σημαίνει ότι δεν μπορεί να αφήσουμε απ' έξω την ε, Κίνα, ιδίω για τον κλάδο του ίνου που είναι ε, η καραμέλα για να ανοίξει το δρόμο. Με το, κρασί, με το, το κρασί ανοίγει τα σύνορα και μετά μπαίνουν άλλες, ε, άλλα προϊόντα στις τρίτες χώρες. Να συγχαρώ λοιπόν ε, την Επιτροπή μας για την ερώτηση αυτή και ελπίζω να γίνει η συζήτηση στην Ολομέλεια το συντομότερο δυνατόν για να μπορέσω να μετάσχω σε αυτήν και να δει ο κλάδος ότι το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται σοβαρά για τα προβλήματα του αμπελοϊνικού κλάδου. Ο κ. Βόλφκαν από την Επιτροπή. welcome. We love to listen to the Commission. Θα θέλαμε να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. functioning So, <clears throat> So we have Εδώ δουλεύει το μικρόφωνο. Ένα πρόβλημα το λύσαμε. Πρώτα πρώτα να πω ότι ο Επίτροπος δεν έχει πρόβλημα να σας απαντήσει στο ερώτημα αυτό και ευχαριστώ που δίνετε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το λόγο και δεν έχουμε πρόβλημα να απαντήσουμε και σε άλλες τεχνικές ερωτήσεις ενδεχομένω για το ίδιο θέμα. Λοιπόν, πρώτα πρώτα ελέγχθη ότι εδώ και εδώ πρόκειται για μέτρο ουσιαστικά αντιπίνων, ανταποδοτικά μέτρα. Ε. Κάθε μέλος του ΠΟΕ έχει δικαίωμα να εφαρμόσει τέτοιου είδους μέτρα εάν συντρέχουν κάποιες νομικές προϋποθέσεις, περιστάσεις και από νομικής απόψεως λοιπόν μπορεί να το κάνουν όλοι αυτοί, αυτό όλα τα μέλη του ΠΟΕ. Είναι νόμιμο το να πάρει κανείς τέτοια μέτρα ε, βέβαια γίνονται κάποιες ε, έρευνες, ε, εμείς ε, συμμετέχουμε στην έρευνα που γίνεται ε, μαζί με τα κράτη-μέλη και την Κομισιόν. Η Κομισιόν δουλεύει πολύ στενά με τα τρία κράτη-μέλη τα οποία εμπλέκονται και κάποιους εθνικές ενώσεις εινοπαραγωγών και τα για να προχωρήσει η υπόθεση με τον καλύτερο τρόπο. Ο Επίτροπος Τεχούχτ συμφώνησε και με τον κύριο Κάου ότι θα υπάρξει και διάλογος business to business για να διευκολυνθεί η επίλυση του θέματος και πράγματι και εκείνα να υποσχέθηκε ότι κατά τη διάρκεια του διαλόγου δεν θα εφαρμοστούν τα ανταποδοτικά μέτρα τα μέσα Απριλίου είναι η επόμενη συνάντηση για το διάλογο αυτό. Έχετε το υπόψη σας και νομίζω ότι εδώ μπορώ να κλείσω αλλά σας διαβεβαιώ ότι η Κομισιόν ε, καταβάλει πάσα προσπάθεια για να υποστηρίξει τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού αμπελοϊνικού τομέα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Το κείμενο της προφορικής ερώτησης ε, το έχετε όλοι, θα ψηφίσουμε αύριο και η ολομέλεια στην οποία θα γίνει η επόμενη ψηφοφορία δεν είναι ακόμη καθορισμένη, μπορεί να είναι Φεβρουάριος, μπορεί να είναι Μάρτιος. Προχωρώ στο σημείο 7. Αποστολή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Ε, ξέρουμε πολλά πράγματα που μας τα είπε ο κύριος Μιταράκης. Ε, πιο παλιά η αντιπροσωπεία αυτή ήταν ε, ολιγομελής συναντηθήκαμε με προσώπους της κυβέρνησης, της Βουλής, των επιχειρήσεων, των συνδικάτων και επισκεφθήκαμε και μια πολύ καινοτόμα εταιρεία καλλιντικών που είναι κοντά στην Αθήνα. Ακούσατε το κύριο Μηταράκη μας ανέφερε τους στόχους και τις δεσμεύσεις της ελληνικής προεδρίας στον τομέα του εμπορίου. Θεωρούμε ότι οι φιλοδοξίες είναι μάλλον ρεαλιστικές. Βεβαίως ο χρόνος που έχει στη διάθεσή της η, η ελληνική προεδρία δεν είναι και πολλής διότι θα γίνουν και εκλογές το Μάιο στην Αθήνα είπα αυτό που είπα και σήμερα εδώ ότι αν θέλουμε να επιτύχουμε οτιδήποτε για τα θέματα αυτά θα πρέπει να είμαστε αρκετά σκληροί με το Συμβούλιο πρέπει να υπάρχει και βούληση να κάνουμε παραχωρήσεις και εμείς αλλά και οι άλλοι και το Συμβούλιο πρέπει να κάνει κάποιες υποχωρήσεις. Εδώ τα πράγματα είναι αμοιβαία, δεν είναι μονόδρομος. Η υπόθεση και η ΜΕΝ και η ΔΕ και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα πρέπει να κάνουν προσπάθειες. Λοιπόν, δεν ξέρω, κύριε Καζάκ, έχετε σχόλια ή... Όχι ακριβώς, πρόεδρε, νομίζω ότι αυτά που είπατε είναι ορθά. Εγώ ζήτησα το λόγο μονάχα για να πω ότι με εντυπωσίασε ο ενθουσιασμός και η φιλοδοξία πραγματικά της ελληνικής προεδρίας η οποία μέσα στον πολύ σύντομο χρόνο που έχει στη διάθεσή της θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Βεβαίως όπως είπατε πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να μην έχουμε υπερβολικές προσδοκίες αλλά αν συνεχίσουμε να δρούμε σε στενή συνεργασία με το Συμβούλιο νομίζω ότι πολλά μπορούμε να επιτύχουμε. Ζητώ λοιπόν να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία με το Συμβούλιο Σίγουρα θα υπάρξουν προβλήματα στην επίλυση ορισμένων θεμάτων, ιδιαίτερα νομοθετικών θεμάτων, αλλά θα πρέπει να συνεχιστεί η συνεργασία για να επιτύχουμε ό,τι μπορούμε. Πρόεδρος, να πω και κάτι τι, όταν είμαστε... Όταν είμαστε στην Αθήνα, ο εκπρόσωπος της Ελλάδας στο TPC σκοτώθηκε σε τροχαίο ατύχημα ε, και ε, γι' αυτό δεν ε, μπορέσαμε να συζητήσουμε πολλά πράγματα. country at the Και, ναι, αλλά πιστεύω ότι μπορούμε ε, να έχουμε εμπιστοσύνη στην κυρία που είδατε σήμερα εδώ και η οποία ε, θα καταβάλει προσπάθειες για να επιτευθούν οι συμβιβασμοί που μας χρειάζονται. Καταλαβαίνετε ότι δεν τα ξέρει και τα θέματα η κυρία είναι καινούργια στο πόστο αυτό. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι ε, φαίνεται ότι πήγαμε πολύ γρήγορα. Θα κάνουμε διάλειμμα λοιπόν μέχρι τις 5.30 όπου θα συνεδριάσουν, οπότε συνεδριάσουν οι συντονιστές. Έτσι. Μόνο ο Σόλτσο ε, είναι εδώ από τους συντονιστές βλέπω. Οι υπόλοιποι μπορείτε να φύγετε. Γεια σας και θα τα ξαναπούμε αύριο το πρωί. Περιμένουμε όμως τους συντονιστές που ελπίζουμε ότι θα έρθουν όλοι τους.